I think we can start. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ja, liebe Kolleginnen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της σημερινής μας συνεδρίας. Να σας ε, συστήσω τον Μάρκ Καλοσιέση, που είναι ο νέος μας συνάδελφος στη γραμματεία της Επιτροπής Τραν. Καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Η μερίσια διάταξη εγκρίνεται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι από ό,τι βλέπω. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Τέταρτο θέμα. Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Κύρκο, για να μας ε, παρουσιάσει σύντομα την γνωμοδότηση του. Κύριε Κύρκο, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chair. I will speak in Αγαπητοί συνάδελφοι, τον Ιούλιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Συμβουλίου να αναλάβει την ανάλυση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει στην ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης για την πολιτιστική κληρονομιά. Εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αναλάβαμε να προσεγγίσουμε τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα διακυβεύματα που δημιουργούνται από τις συνέργειες μεταξύ του πολιτισμού και του τουρισμού. Με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού εισηγείται στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία, που είναι επί τη ουσία αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα, να συμπεριλάβει προτάσει για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Όπω γνωρίζετε, η Ευρώπη είναι ένα από του σημαντικότερου πολιτιστικού τουριστικού προορισμού στον κόσμο. Ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, μέσα από την αυθεντικότητα και την πολυμορφία της, αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημά της στον τομέα του τουρισμού και αναπόσπαστο μέρος της ανταγωνιστικός της. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε ώστε να παραμείνει η Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Ο πολιτιστικός τουρισμός, που είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, συμβάλλει λοιπόν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό τονίστηκε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Τουρισμό που πραγματοποιήθηκε στην Άπολη τον Οκτώβριο. Επίση, συμβάλλει στη μείωση του εποχικού και γεωγραφικού συγκεντρωτισμού του προσφερόμενου προϊόντο. Ο πολιτιστικό τουρισμό δημιουργεί ευκαιρίε για την ανάπτυξη τη επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό από μικρομεσαίε επιχειρήσει που ενεργοποιούνται στον χώρο αυτό, το 95% των επιχειρήσεων του τομέα. Είναι σημαντικό λοιπόν να στηρίξουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη διατήρηση, προστασία και προώθηση της πολιτικής κληρονομιάς μας. Κλειδί για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και η υψηλού επίπεδου επαγγελματικές δεξιότητες. Η Ευρώπη θα πρέπει να διευκολύνει την πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων για τα διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τον πολιστικό τουρισμό. Ο αποτελεσματικό σχεδιασμό και η διαχείριση τη τουριστική ανάπτυξη προποθέτει τη σύμπλευση των υπευθύνων χάραξη πολιτικής με τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες και τα δίκτυα των τουριστικών πρακτόρων. Ζητούμε από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να δρομολογήσουν έναν πανευρωπαϊκό διάλογο μεταξύ τους και να στηρίξουν τις συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και των συναφών ΜΚΟ σημαντικό ρόλο για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων έχουν οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υποστηρίζουμε την Επιτροπή στις πρωτοβουλίες αυτές. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί επίσης μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για την τοπική ανάπτυξη. Χωρί να αμφισβητείται η σημασία του αστικού τουρισμού, τονίζουμε ότι πολιτισμό προσφέρουν και οι αγροτικέ και νησιωτικέ περιοχές με λαϊκή τέχνη, βιοτεχνία, λαογραφία, χειροποίητα, γαστρονομικές παραδόσεις, τα τοπικά προϊόντα και φεστιβάλ, το άθικτο φυσικό περιβάλλον. Για να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα των μικρότερων και των απομακρυσμένων αυτών τουριστικών προορισμών και να αναδειχθεί ο πλούτος τους, είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τι πολυτροπικέ διασυνδέσει. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαπεριφερειακή και διασυνοριακή ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων. Τα διεθνικά πολιτικά, πολιτιστικά τουριστικά προϊόντα αντικατοπτρίζουν τις κοινέ ευρωπαϊκές μας αξίες. Παράδειγμα διακρατικών πανευρωπαϊκών θεματικών για τον τουρισμό που βασίζεται στην κοινή πολιτιστική ταυτότητα μιας ευρύτερης περιοχής αποτελούν φυσικά οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές τις οποίες προωθεί η Επιτροπή σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στηρίζουμε τη συνέχιση της χρηματοδότησής του. Δεν ξεχνούμε τι ήδη πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε που αξιοποιούν την κοινή κληρονομιά της Ευρώπης με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως οι ευρωπαϊκέ ποδηλατικέ Διαδρομές, οι πολιτιστικέ Πρωτεύουσες της Ευρώπης, το δίκτυο Europa Nostra, το δίκτυο Natura 2000, το Σήμα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, οι Ευρωπαϊκέ ημέρε Πολιτιστική Κληρονομιά κτλ. Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή μου τονίζοντα ότι η διασφάλιση τη συνέργεια τουρισμού και πολιτισμού θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική όμω για τη σωστή και οικονομική σύζευξη πολιτισμού και τουρισμού θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό στην ηθική και συμβολική αξία των πολιστικών μνημείων και στην προστασία και διατήρηση τόσο αυτών όσο και του περιβάλλοντος τοπίου της τοπικής κουλτούρας. Είναι ζωτική σημασία οι πολιτικέ για το τουρισμό να βασίζονται στον βιώσιμο, υπεύθυνο και ποιοτικό τουρισμό και να μπορέσουν να αποτρέψουν τι ενδεχόμενε αρνητικέ επιπτώσει του μαζικού τουρισμού και να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την πολυμορφία των τοπικών πολιτισμών. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Γραμματεία τη Επιτροπή Μεταφορών και του πολιτικού συμβούλου τη ομάδα μου για την πολύ καλή συνεργασία. Ευελπιστώ σε μια καλή συνεργασία και με τους κοιόδη εισηγητέ, με τους οποίους οργανώνεται συνάντηση τις προσεχής μέρες, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους, προκειμένου να εμπλωτιστεί το κείμενο και με τις δικέ τους πολύτιμε ιδέες και προτάσει. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Ο κόσμος Λωτός έχει το λόγο πρώτος. Ένα λεπτό. Λέει ο πρόεδρος. Επειδή δεν είναι εδώ η σκιώδης του ΕΛΚ, θα ήθελα να μιλήσει ο κύριος Βιμ, Βαντεκάμπ. Eh, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η κυρία Σουίτσα, δεν είναι εδώ, ε, πρέπει να το είχα πει από πριν, ε, είναι απούσα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή εκ μέρου του ΕΛΚ για αυτή την πολύ σαφή έκθεση την οποία μας παρουσίασε. Η σημασία στην σύνδεση ανάμεσα στον τουρισμό και τις μεταφορές είναι προφανής. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά σε γενικές γραμμές η έκθεση μας ικανοποιεί. Σας ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριο Λοτόφσκι τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ορισμένα λόγια εκ μέρους του Τόμας Πορέμπα που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Θα το κάνω στα πολωνικά όμως, αν μου επιτρέπετε. E, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, εισηγητή για αυτό το προσχέδιο και ιδιαίτερος για το γεγονός ότι ε, υπογράμμισε ε, θέματα όπως το, ο ποδηλατικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός προσκυνήματος κλπ. Ε, επίσης υπάρχει και το, η δυνατότητα ε, διαδρομής ε, του σιδηρού παραπετάσματος. Είναι ένα project το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την πολιτική μας κληρονομιά. Πρόκειται για 9.000 χιλιόμετρα, μια διαδρομή 9.000 χιλιόμετρων μέσα από πολλά κράτη-μέλη από την, ε, ε, και βέβαια μέσω της ε, Ρωσίας, της Γερμανίας, τελειώνει στην Βουλγαρία. Πρόκειται για εκατοντάδες χρόνια ιστορία μας. Μετά από 70 χρόνια μετά τη Σύνοδο της Γιάλτας είναι επίκαιρο. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Τώρα, ε, οι διαδρομές προσκυνήματος και θρησκευτικού τουρισμού και πάλι πρόκειται για την ευρωπαϊκή κουλτούρα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές κοινότητες. Στην Πολωνία έχουμε 500 ε, σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ε, ναούς και άλλα, η πρόσβαση σε αυτά εξαρτάται κατά πολύ από την δυνατότητα ε, ε, να φτάσει κάποιος με τα μέσα μεταφοράς κλπ. Ο πολιτιστικός τουρισμός έχει σχέση προφανώς με επίσκεψη σε σημεία ενδιαφέροντος όπως μουσεία και άλλα. Ε, αυτές οι επισκέψεις συνήθω αποτελούν τμήμα ε, πακέτων, τουριστικών πακέτων. Ο πολιστικός λοιπόν ε, τουρισμός ε, θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη πρόσβαση και εύκολη πρόσβαση γιατί αλλιώς μεν τουρίστες θα ε, κάνουν πίσω. Χρειάζεται λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια εύκολη πρόσβαση σε όλα αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα να, να τα προωθήσουμε όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ε, η πρόσβαση ε, άλλωστε σε τέτοιου είδου μνημεία μπορεί να βοηθήσει και στην καλύτερη αλληλοκατανόηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τους φιλελεύθερους. Ο Παύλ Τέλτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το συγγνώμη από τον συνάδελφο διότι ο Πάβελ παραδίδει κάποια έκθεση σε κάτι παρόμοιο στην Οικονομική Επιτροπή οπότε θα πω μερικά λόγια εκ μέρους της συναδέλφου. Όπως ακούτε η φωνή μου δεν είναι και σε πολύ καλό επίπεδο σήμερα. Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι πολύ σύντομος. Να προσθέσω ίσως ένα-δύο δικά μου στοιχεία. Θα είμαι τάχιστος. Πρώτα απ' όλα εκ μέρους της Μαρτίνα εκτιμώ και εγώ την έκθεση Πιστεύω ότι είναι πολύ καλά σταθμισμένη, πολύ καλά εστιασμένη, ισορροπημένη έκθεση. Η Μαρτίνα δεν αποκλεί να έχει μία-δύο τροπολογίες, αλλά βασικά υπάρχει ευρεία συμφωνία με αυτά που συμπεριλάβατε στην έκθεσή σας και την όλη αντίληψη και προσέγγιση που ακολουθήσατε. Να προσθέσω ίσως κάποια ίσονο σημασία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, δίνεται έμφαση στη διατροπική μεταφορά αλλά στα πλαίσια ε, των πλέον απομακρυσμένων περιοχών και μόνο. Και νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά προϋποθέσεις για τόνωση του τουρισμού, του πολιτισμικού, να τα πάρουμε όλα μαζί. Αυτή η διατροπικότητα είτε είναι για πομακρισμένες περιοχές ή μικρές περιοχές να ληφθούν υπόψη. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, και αργότερα στο έτος θα δούμε κάποιε πρωτοβουλίε για τα εισιτήρια και τις κρατήσεις κλπ. Και κάτι άλλο που έχω να πω. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κρισίμου σημασίας και στον τουρισμό. Και θα το εκτιμούσαμε αν γινόταν μνήα της ανάγκης να καλύψουμε τη δυσανάλογο, το δυσανάλογο διοικητικό άχθος, το, το υπερβολικά ρυθμιστικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν καμιά φορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως μια τέτοια αναφορά θα ήταν καλή, θα ήταν ευπρόσδεκτη. Θα βοηθούσε να τονώσουμε τις επιχειρήσεις και ίσως να ενθαρρύνουμε κάποιους να ασχοληθούν με τέτοιες επιχειρήσεις. Τελευταίο σχόλιο. Στα πλαίσια του σημείου 9 ε, ίσως εκεί μπορούμε να αναφέρουμε την ευρωπαϊκή ε, πρωτεύουσα της ε, νεολαίας, της νεότητας. Ευχαριστώ. Γκούε, Μέγια ή κάποιος άλλος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαίρετη δουλειά του εισηγητή Το, έχουμε, το σκεφτόμαστε εδώ και αρκετό καιρό για το πώς θα μπορούσαμε να ε, αξιοποιήσουμε την τόσο πλούσια ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά ε, σε συνδυασμό με τον τουρισμό. Πώς θα μπορούσαμε να την προβάλλουμε μέσω του τουρισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Στο πλαίσιο αυτού λοιπόν του προβληματισμού ε, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τα δίκτυα μεταφορών και θα πρέπει στην Ευρώπη να σταθμίσουμε το ενδεχόμενο ε, να πάρουμε ως κριτήριο την ανάπτυξη των ε, μεταφορικών, των δικτύων μεταφορών ε, για την προβολή του, της πολιτικής οικονομίας. Δηλαδή να μην έχουμε τρία ανεξάρτητα στοιχεία, τα, η κληρονομιά, και ο τουρισμός θα πρέπει να ειδωθούν ως τμήματα της ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Εύανς. Κυρία Εύανς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ε, καλά ισορροπημένη γνωμοδότηση Θέλω και εγώ να συμφωνήσω με, την, ε, ε, με τον τονισμό της σημασίας του τοπικού τουρισμού και του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει ε, σχέση μεταξύ της διατήρησης του, της πολιτικής κοινωνίας και του τουρισμού. Μπορούν να αποτελέσουν, ο τουρισμός μπορεί να τονώσει ε, μια περιφέρεια γιατί ακριβώς μπορεί να αναδείξει η περιφέρεια αυτά ε, τι, έχει να προσφέρει σε τουρίστες αλλά ταυτόχρονα μπορεί να παράσχει μια πλατφόρμα και για τους, ε, το, τους κατοίκους της περιοχής για να γνωρίσουν καλύτερα την ίδια τους περιοχή Γι' αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται στην γνωμοδότηση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ίσως να κάνουμε κάποιες αλλαγές για να τονιστεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι η επιτυχία του τουρισμού εξαρτάται πραγματικά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά υπάρχει και το θέμα της εποχικότητας, ε, κάτι με το, το οποίο είχαμε συζητήσει και με την Κομισιόν ε, στην συζήτηση που είχαμε κάνει για τον τουρισμό πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί λοιπόν ε, αυτός ο στόχος μέσω των μικρομισίων επιχειρήσεων και ο υπεύθυνο ε, τουρισμός επίσης εξαρτάται από αυτές. Ένα άλλο θέμα που δεν είδα να συμπεριλαμβάνεται είναι ο ρόλος των γλωσσών στην πολιτιστική κληρονομιά και στον τουρισμό και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι προφανές ε, είτε πρόκειται για επίσημη γλώσσα της Ένωσης ε, είτε για γλώσσα ε, μικρής εμβέλειας μπορούν όλες αυτές οι γλώσσες να αποτελέσουν παράθυρο για την πρόσβαση των ανθρώπων στον πολιτισμό. Οπότε νομίζω ότι και τις γλώσσες δεν θα πρέπει να τις ξεχάσουμε γιατί αποτελούν σημαντικό παράγοντα κατανόησης της ιστορίας και των χαρακτηριστικών μιας περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τζέκι Φώστερς. Η Τζάκη Φώστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ο τουρισμός πράγματι ήταν μια σταχτοπούτα. Αν δούμε όλα όσα συζητήσαμε επί σειρά ετών. Και σωστό είναι αυτό που είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Δηλαδή πόσο σημαντική είναι η αλυσίδα εφοδιασμού και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που περνούν από μεταφορά στον τουρισμό. Και δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στην Ευρώπη ε, δημιουργούνται στα πλαίσια του τουρισμού είναι καλό να τίθεται τα θέματα, να τονίζουμε το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να πω κάτι. Μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά. Εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ ακριβά παλαιά κτίρια. Πολύ δύσκολο και είναι ακριβά να συντηρηθούν. Και πρέπει να εξισορροπηθεί και με τον τουρισμό και αν θα πρέπει να πληρώνουν οι τουρίστες κλπ. Αυτό είναι ευθύνη των ε, κρατών μελών. Και δεν θέλουμε να δούμε κάτι που αφαιρεί την ευθύνη του κράτους μέλους να έχει μια σωστή τουριστική βιομηχανία. Και να θεωρεί το κράτος ότι θα δίνει διάφορα χύψη ωμέγα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνει αυτό. Διότι πρέπει να το ρυθμίσει η χώρα. Βέβαια, συνεργασία είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει. Μπορούμε να προσφέρουμε πολλά στη μεγάλη αυτή ήπειρο τη Ευρώπης και δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα πήγαινε, θα πήγαινε οπουδήποτε αλλού τη Ευρώπη. Δομινίκ Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Το κείμενο είναι πολύ πυκνό και πλούσιο να κάνω συμπληρωματικά σχόλια. Πρώτο, η κρίση η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έπληξε πολύ σοβαρά τον πολιτισμικό τομέα στην ε, Ευρώπη. Δεύτερη παρατήρηση. Ίσως θα μπορούσαμε πούμε σαφέστερα στην έκθεση την ηλική κληρονομιά, κάτι που αναφέρθηκε από πολλούς παρεμβαίνοντες, και την άειλη κληρονομιά που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και μεγάλος παράγοντας τουριστικής ελκυστικότητας Μιλήσαμε πολύ για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν. Να υπογραμμίσω και το εξή. Ότι στην Ευρώπη ε, συχνά δεν είναι εμπορική φύση. Είναι στα χέρια ενώσεων ε, διαφόρων ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών ε, ιδρυμάτων κλπ. Και αυτές, αυτές υπέφεραν, οι φορείς υπέφεραν πάρα πολύ διότι λόγω της οικονομικής κρίσης περιεκόπησαν οι πόροι που είχαν. Εξ αυτού και είναι συμπληρωματική σκέψη, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του αντιχτύπου που έχει η κρίση στον τομέα το πολιτισμικό, μεταξύ των χωρών της ανταγωνιστικότητας που ε, έχουν διαρθρωμένη προσέγγιση για την πολιτισμική ε, κληρονομιά είτε σε εθνικό επίπεδο όπως η Γαλλία είτε ιδιωτική πολιτική, κίνητρα φορολογικά, ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις χώρες της συνοχής όμως δεν υπάρχει διαθροτική υποστήριξη που να είναι σταθερή για τις πολιτισμικές δραστηριότητες. Και όσα είναι εκτός του εμπορικού συστήματος επλήγησαν πολύ από την κρίση και αυτό είχε και αντίκτυπο και στις εμπορικές δραστηριότητες. Αν έχετε θειάσους, χορού, θεάτρου ή μουσική εμπορικά συγκροτήματα ε, που είναι μη εμπορικής φύσεως καταραίουν τελικά λόγω της ε, οικονομικής κρίσης αυτές οι δραστηριότητές τους. Κάτι που ανέφερε η έκθεση σωστά. Υπάρχει κάποια διαφορά, κάποια αντίθεση αν θέλετε, μεταξύ των εξή. Ο τουρισμός είναι 8,5% του ΑΕΠ της Ενώσεως το μισό του ΑΕΠ εξαρτάται από δραστηριότητες άειλες ή υλικέ πολιτισμικές. Ας μιλήσουμε για το 7% του ΑΕΠ της Ένωσης που εξαρτάται από ένα τομέα που έχει πληγεί τα μάλα από την κρίση και δεν έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης ε, από, από την πλευρά μας. Εμείς μιλάμε για τον τουρισμό και έχουμε τα μέσα που ξέρετε, μηδέν. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη ασχολείται από τον πολιτισμό έχει οικονομικά μέσα ε, πολύ περιορισμένα. Άρα υπάρχει αντίθεση μεταξύ ενός πολύ δυναμικού τομέα, ενός τομέα που είναι σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ, που αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της ε, διαθροτικής μορφής και της ανομοιογένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και απ' την άλλη έχουμε την αδυναμία υποστήριξης ε, από πλευράς των πολιτικών θεσμών, είτε εθνικών είτε ευρωπαϊκών. Θα ήταν ενδιαφέρον να υπογραμμίσουμε παρόλα αυτά τον εύθραυστο χαρακτήρα και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει αυτός ο τομέας. Όσον αφορά τη Γαλλία, 25% των αήλων πολιτικών θεσμών εξαφανίζονται. Και βέβαια αυτό δεν είναι ότι αφήνει και τον τουρισμό εν γέννη χωρίς να δημιουργεί συνέπειες για αυτόν. Ευχαριστώ κύριε Όλγα Σελένοβα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική γνωμοδότηση, πολύ ισορροπημένη. Περιγράφει και τους κινδύνους προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Δυο σχόλια. Πρώτον, το σημείο 8 της έκθεσης. Χαίρομαι που αναγνωρίζεται η σημασία των διαπεριφερειακών ε, δραστηριοτήτων. Όμως θα πρέπει να μιλήσουμε και για την απόσυρση των φραγμών που υπάρχουν, κατάρριξη των φραγμών για τις διασυνοριακές μεταφορές. Για παράδειγμα θα πρέπει να έχουμε ε, διεθνή τιμολόγηση για τις συνδρομικές μεταφορές. Ε, αυτή τη στιγμή, περνώντας τα σύνορα, μπορούμε να βρούμε ε, τιμές ε, σιδηροδρομικές, ε, για σιδηροδρομικές μεταφορές 7 με 9 φορές ακριβότερες ή φτηνότερες αντίστοιχα. Ε, για παράδειγμα, τα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Αυστρίας. Μετά, βιώσιμος τουρισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε την σημασία των υποδομών που θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, Τέντρα Κλούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση αυτής της ε, γνωμοδότησης και νομίζω ότι η ε, απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και αυτό ε, αφορά, ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι το 40% του τουρισμού προέρχεται από τρίτες χώρες και αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, για την κουζίνα, για τις γλώσσες, για όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση αυτή και Σημαντικό είναι ότι γίνεται έκκληση προς την Κομισιόν ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν για τη διατήρηση, τη διαφύλαξη της πολιτικής κληρονομιάς και νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να αυξήσουμε αυτό το 40%. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Ε, υπάρχει και ε, έκκληση να διευκολύνει η Κομισιόν ε, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τη διατήρηση, τη διαφύλαξη της πολιτικής κληρονομιάς και εγώ νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ από προσωπική μου εμπειρία μπορώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη από το ευρωπαϊκό επίπεδο σε, αυτό τον, σε, αυτούς τους φορείς για να υπάρχει διατήρηση, διαφύλαξη της πολιτικής κληρονομιάς. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι ανάγκη να τονίσω εγώ πόσο σημαντικό είναι για μένα προσωπικά το θέμα, αφού ε, και εγώ ο, ο ίδιος θέτω το ζήτημα αυτό πολύ συχνά. Συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες και δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχουν ήδη ακουστεί. Αλλά να προσθέσω το εξή. Τι τελευταίε δεκαετίε άλλαξε ο χαρακτήρα του τουρισμού παγκοσμίω. Στην Ευρώπη έχουμε τουριστικά ισχυρέ χώρε, όπω για παράδειγμα η Ιταλία, η Γερμανία η οποία επίσης προσελκύει πολλούς τουρίστες. Θα μπορούσα να αναφέρω και τη Βουδαπέστη που είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη. Ωστόσο υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο και αυτό είναι η παγκόσμια αλλαγή στον τομέα του τουρισμού. Ένας τουρίστας από τις ΗΠΑ ή από κάποια αραβική χώρα επισκέπτεται πλέον περισσότερους από έναν προορισμού στην Ευρώπη. Στις ε, διαφημίσεις, αν δείτε, υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα προορισμών ε, από το οποίο μπορεί κανείς ε, να επιλέξει Ντουμπάι, Μεξικό, Νότια Αμερική. Αυτό που για μας στην Ευρώπη είναι χαρακτηριστικό και το οποίο δεν μπορεί να το ε, ανταγωνιστεί και ο υπόλοιπος κόσμος είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Διότι αυτά που έχουμε εμείς εδώ στη γυραιά Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να το χτίσει κανείς, να το αντιγράψει κανείς ούτε στο Ντουμπάι ούτε στην Ασία. Είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Η ευρωπαϊκή πολιτιστική μας κληρονομιά. Και αυτό είναι το κύριο σημείο που νομίζουμε, νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε, δηλαδή να αποτελέσει εμάς, για εμάς αυτό το, το, το μήνυμα προς την Κομισιόν και προς τα Εθνικά Κοινοβούλια, ότι βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά έντονο ανταγωνισμό και εμείς έχουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Εδώ δεν μιλάμε για επενδύσεις, για χρήματα. Μιλάμε για το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημά μας αυτό στον κόσμο, στον κλάδο του τουρισμού. Το αν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, το αν θα μπορέσουμε να εξεύρουμε τους πόρους για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη τις επόμενες δεκαετίες, είναι και αυτά στοιχεία που θα ήθελα να τα θέσω έτσι εδώ στη συζήτηση. Την Πέμπτη θα συμμετάσχω σε ένα, ε, συμμετείχα, με συγχωρείτε, σε ένα συνέδριο στην Μαδρίτη όπου τονίστηκε και από την πλευρά του ΟΗΕ ότι ο πολιτιστικός, κληρονομιάς, ο, πολιτιστικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός. Να ξαναευχαριστήσω και εγώ τον ε, εισηγητή. Πρόεδρος, ε, επειδή αναφέρθηκε το σιδρούν παραπέτασμα, θα ήθελα να πω τα εξή. Ιστορία και πολιτισμός είναι δύο πράγματα που δεν, μπορούν να, δεν μπορεί να τα διαχωρίσει κανείς. Στο Βερολίνο την πόλη καταγωγής μου, έχει μετρηθεί ότι το 80% ε, των τουριστών έρχονται λόγω της ιστορίας της πόλης. Κάτι τέτοιο μπορούσε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της διαδρομής για το σιδηρού παραπέτασμα. Υπάρχει βεβαίως και η επέτειος της Συνόδου της ε, Γιάλτα, του τέλους του ε, Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, Παγκοσμίου Πολέμου και ε, του χρόνου θα έχουμε και την 25η επέτειο της ανεξαρτησίας των βαλτικών χωρών. Πρόκειται για πολιτισμό και ιστορία ταυτόχρονα. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην ε, Κλαϊμπέντα υπάρχει ε, ένα ε, συντριβάνι που υπάρχει και ένα μικρό παπάκι, υπάρχει και ένα ωραίο παιδικό τραγουδάκι στα γερμανικά όλη αυτή η περιοχή ε, είχε κάποτε είχε διάφορες, ε, ε, υπήρχαν διάφορα σύμβολα παλιά υπήρχε ένα παπάκι στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από ένα κόκκινο αστέρι και τώρα ξανά υπάρχει ένα παπάκι επίσης το σιδρού παραπέτασμα περνά παράλληλα με την λεγόμενη πράσινη ζώνη, το Green Belt στην ε, ε, ζώνη αυτή, ε, η ζώνη αυτή είναι στην ουσία μια ζώνη φυσικής ανάπτυξης φυτών. Υπάρχουν φυτά και ζώα σε αυτή τη ζώνη όπου υπήρχε παλιά το σιδούν παραπέτασμα που είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Γι' αυτό ε, το λόγο φαίνεται ότι ε, όλα αυτά βεβαίως ε, έχουν είναι σημαντικά από οικολογική, ιστορική, οικονομική άποψη για ε, χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό. Οπότε αυτέ τι χώρε θα πρέπει να τι βοηθήσουμε και στον τομέα του πολιτισμού. γι' αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή εκτός από τον τουρισμό και στον πολιτισμό. Ε, ο εισηγητής έχει τον λόγο αν θέλει για μια τελευταία φορά. Alles ist gesagt. Dann bedanke ich mich. Ωραία. Τότε. This discussion in more θα περιμένουμε την συνέντευξη τη επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε πιο πρακτικά τις συγκεκριμένε τροπολογίε. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Προθεσμία είναι 13 Μαρτίου 2015 για την υποβολή των τροπολογιών στις 15 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι. Ε, θέμα 5. Παρουσίαση της Κομισιόν από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ για τη θαλάσσια επιτήρηση. Θα ήθελα αρχικά να δώσω τον λόγο στην Παρατεγμίντα ε, από την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε λίγο εδώ το πώς καθόμαστε πάνω στο βήμα. Θα τα καταφέρουμε όμως.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 Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε σας σήμερα. Με ενδιαφέρον άκουσα την παρατήρησή σας, διότι και το δικό μου τμήμα εξετάζει τις, ε, ε, ε, το, την πολιτική οικονομία που βρίσκεται στη θάλασσα, υποθαλάσσια. είναι και αυτό σημαντικό, αλλά σήμερα θα σας μιλήσω για την ε, θαλάσσια επιτήρηση. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που υιοθετήσαμε πέρσι και θέλουμε να τη συζητήσουμε μαζί σας. Έχουμε ήδη παρουσιάσει την ε, μπλε ανάπτυξη, τη γαλάζια ανάπτυξη για την ε, ε, την ολοκλήρωση των, της, ε, των πολιτικών για τη θάλασσα. Εστιαζόμαστε πλέον στην γαλάζια οικονομία και στη γαλάζια ανάπτυξη ε, μέσω ενοποίησης κλάδων που θα επιτρέψουν βιώσιμη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα επιτρέψουν επίσης να χρησιμοποιούμε την θάλασσα ως καλύτερο τρόπο για τη δημιουργία μιας ολόκληρης αλυσίδας ε, προσθέμενης αξίας από την στεριά στη θάλασσα. Έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένου ε, τομείς οι οποίοι θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα ε, και που είναι ατμομηχανές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην γαλάζια οικονομία. Για παράδειγμα μεταφορές, ναυπηγική, ξορυκτική βιομηχανία στη θάλασσα κλπ η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει όλη αυτή την ατζέντα ε, για την απασχόληση ε, αλλά ε, και για οικολογικούς λόγους. Θέλουμε συνεργασίες σε πλαίσιο μακροπεφιακών στρατηγικών με συνολικές και εστιασμένες στρατηγικές και εργαλεία. Λυπάμαι πολύ, το PowerPoint μου δεν με ακολουθεί. ωραία. Όλα αυτά τα εργαλεία, οριζόντια εργαλεία ε, που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εμπλέκουν πολλούς τομείς και, ε, πολλούς, ε, και πολλές οντότητες οι οποίοι θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα σύστημα επιτήρησης, θαλασσής επιτήρησης. Έχουμε 400 αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που παρατηρούν και επιτηρούν την ε, θάλασσα. Ραντάρ, ε, πλοία, αεροσκάφη, συστήματα πληροφοριών, δορυφόροι κλπ. Σε 7 θαλάσσιους τομείς. Έχουμε επιθεωρήσεις μεταφορών, περιβαλλοντικές, επιθεωρήσεις στην αλληλεία, στα σύνορα, στα τελωνία, την δυνάμεις της επιβολής της τάξης και βέβαια στην ε, άμυνα. Έχουμε λοιπόν πολλές πληροφορίες που συλλέγονται από όλους αυτούς τους φορείς, από όλες αυτές τις οντότητες ε, και που κάθε μία έχουν συγκεκριμένες, έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες ε, στο θέμα της ακτοφυλακής κλπ. Έχουμε πολλές ε, πηγές πληροφοριών, από μυστικές πληροφορίες, από επίσημες εκθέσεις, από πλατφόρμες, από βάσεις δεδομένων κλπ. Οπότε πριν από μερικά χρόνια είπαμε έχουμε μια τεράστια ευκαιρία διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων αυτών των ε, φορέων. Και γι' αυτό το λόγο ε, ενδεχομένως θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσα στο πλαίσιο του υπαρχόντος νομικού πλαισίου. Ε, εδώ λοιπόν έχουμε τους, ε, τις διάφορες ε, λειτουργίες, ακτοφυλακή, τις διάφορες επιτηρήσεις, έλεγχο συνόρων, αλληλευτικούς ελέγχους κλπ. κλπ, κλπ. Όλοι αυτοί οι φορείς δημιουργούν πληροφορίες. Το 80% όλων των πληροφοριών αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντοπισμένο σε εθνικά συστήματα πληροφοριών. Όμως 20% των πληροφοριών ήδη την χάνει ανταλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερος μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών, μεταφορών, ε, τη Frontex, δηλαδή του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων κλπ. Θέλουμε λοιπόν αυτό το 20% να το διευρύνουμε και να έχουμε μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και μεταξύ διαφορετικών τομέων και μεταξύ και ε, υπεράνω των συνόρων. κάνουμε μια αξιολόγηση της επιπτώσεων ε, στην ανακοίνωσή μας και είδαμε ότι έχουμε, ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν μέχρι και 17 συστήματα επιτήρησης αλλά που δεν, δεν, λειτουργούν διαλειτουργικά. Ε, όσο πιο ε, μάλλον το ίντερνετ είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να γίνει σημαντική βελτίωση της διαλειτουργικότητας. Ε, είναι μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS, του ασφαλούς πρωτοκόλλου δηλαδή του ίντερνετ, που μπορεί να γίνει αυτός ο διαμερισμός πληροφοριών. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ε, λέμε στην ανακοίνωσή μας ότι μπορούμε να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες που ήδη υπάρχουν και μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών αυτό θα μας αύξανε την επίγνωση της, του ευάλωτου στη θάλασσα, ε, θα μας βοηθούσε να αποφύγουμε ε, τις αλλεπικαλύψεις, θα δημιουργούσε καινούριες υπηρεσίες πληροφοριών και θα βελτίωνε και την συνεργασία μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Συνεπώς ε, έχουμε το, θα μπορούσαμε να ορίσουμε το ε, το περιβάλλον ανταλλαγή πληροφοριών για το θαλάσσιο τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ω μια διαρκή διαδικασία επιθελοντική ε, βάσεω ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Μιλούμε συνεπώς για εθελοντικής φύσεως δραστηριότητα και θα πρέπει να οδηγείται από τις ανάγκες, να έχει ως νόμονα τις ανάγκες και την διάθεση για συνεργασία. Τώρα, ποια θα είναι τα ωφέλη. Θα βελτιώσουμε την επίγνωση των διαφόρων πτυχών ασφάλειας και οικονομικών πτυχών περιβάλλοντος. Θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα, ο συντονισμός των ε, επιχειρήσεων ε, επιτήρησης και θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και την καινοτομία με την δημιουργία καινούριων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, έχουν ήδη αναπτυχθεί πάρα πολλές ε, εφαρμογές. Όλες αυτές οι εφαρμογές είναι σε μεγάλο βαθμό ε, υπηρεσίες πληροφορίας. Ε, αυτό το size λοιπόν θα είναι ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και μια συλλογή από εργαλεία και λύσεις για, την, για να διευκολυνθεί η συνεργασία και η διασύνδεση. Επίσης μια συνεχής διαδικασία για την ε, εφαρμογή δράσεων ε, υπέρ της ε, τεχνικής και λειτουργικής διαλειτουργικότητας. Τι δεν είναι, και αυτό έχει συζητηθεί πολύ, δεν πρόκειται για ένα καινούριο σύστημα επιτήρησης στη θάλασσα, ε, επιτήρησης στη θάλασσα, δεν είναι ένα καινούριο MSA δηλαδή. Αυτό που θέλουμε είναι να ε, συνδέσουμε τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Επίσης δεν πρόκειται για η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, καταχραστεί εθνικών αρμοδιοτήτων. Και τέλος, δεν τελειώνει ε, οποιοδήποτε τύπου τομιακή ευθύνη στον θαλάσσιο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Σε εθελοντικό επίπεδο απλώς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα επίπεδο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Είναι ένα εργαλείο. Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Το έχουμε συμπεριλάβει στο στην ανακοινωσή μας. Έχουμε στους διάφορους τομείς ε, διάφορα νομοθετικά κείμενα, ε, το Safe το ε, Eurosar, κάποια άλλα τα οποία δεν είναι νομοθετικά. Για παράδειγμα το δίκτυο επιτήρησης του ωκεανού, των ωκεανών, ε, το δίκτυο των εθνικών ε, επιτελείο ναυτικού κλπ. Όλα αυτά ήδη υπάρχουν και εμείς δημιουργούμε ένα χάρτη, ένα οδικό χάρτη για την εφαρμογή του ε, συστήματος αυτού, της αυτής που θα ενώνει αυτά τα συστήματα που υπάρχουν ήδη. Ε, θέλουμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ακτοφυλακών. Έχουμε ήδη πιλωτικά προγράμματα στα κράτη-μέλη. Ένα στην Μεσόγειο, το Pumas Med, ένα στη Βαλτική, το Μαρσούνο. Καθένα από αυτά ήταν πιλωτικά με την έννοια ότι θέλαμε να δούμε αν προσθέτουν αξία στην δράση, στις εθνικές δράσεις. Οπότε ε, το 2010 η απάντηση ήταν πως ναι, Υπάρχει προστιθέμενη αξία. Το 2013 ξεκινήσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας ε, για τον εντοπισμό των ε, επιχειρηματικών αναγκών, των επιχειρήσεων δηλαδή. 15 κρατημέλη συμμετείχαν. Ε, έχουμε, είναι το πρόγραμμα EU 2020 ε, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια πλατφόρμα πειραμάτων σε ό,τι αφορά τη Ποιο είναι το πλαίσιο πολιτικής για το ΣΥΖΕ. Ε, πρόκειται για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Το ΣΥΖΕ είναι ένα από τα εργαλεία της. Ταυτόχρονα έχουμε την καινούργια ψηφιακή ατζέντα, ε, την στρατηγική ασφάλεια στην θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΣΥΖΕ βρίσκεται στην τομή αυτών των τριών κύκλων. Ε, αριστερά βλέπετε τον Κάτω αριστερά βλέπετε τον κύκλο της ψηφιακής ατζέντα ε, και της ε, πολιτικής τυποποίησης, η οποία, προτυποποίηση, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για την διαλειτουργικότητα. Ποιες είναι οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το θαλάσσιο ΣΥΖΕ. Θα δημιουργήσουμε ένα εγχειρίδιο ε, πρότυπα διαλειτουργικότητας. Τα κράτη-μέλη θα δημιουργήσουν, ε, θα εξυγχρονίσουν την, ε, τα συστήματα πληροφορικής τους, θα εξασφαλίσουν ότι θα γίνονται σεβαστοί οι κανόνες προστασίας των δεδομένων και θα αναθεωρήσουμε την νομοθεσία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εφαρμογή του θαλάσσιου ΣΥΖΕ. Τι ωφέλη θα προκύψουν από, μια καλύτερη, από ένα καλύτερο διαμοιρασμό των πληροφοριών στον τομέα, στο θαλάσσιο τομέα. Ε, όλοι μαζί θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση της θάλασσας. Ακόμα δεν είχαμε ποτέ ε, σημαντική απειλή τρομοκρατία ή ατύχημα τρομοκρατία στη θάλασσα. Θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό. Θέλουμε να μειώσουμε τους κινδύνου και τι απειλέ και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τη γνώση μας οι πληροφορίε οι οποίε είναι διάσπαρτε στα διάφορα κράτη-μέλη μπορούν να ενωθούν και να μα δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Επίσης αποτελεί στόχο τη ε, στρατηγικής ασφάλειας στη θάλασσα, την οποία εκπονήθηκε πέρσι. με το ΣΥΖΕ θα βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ ε, πολιτικών αρχών αλλά και μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Ε, θα, για παράδειγμα να σας πω Γερμανία. Ε, τα τελωνία και οι συνοριοφύλακες αυτή τη στιγμή κάνουν κοινές, ε, μάλλον ε, χρησιμοποιούν από κοινού τις, τα σκάφη τους και προμηθεύονται από κοινού ο υλικό. Επίσης θα έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, διαφόρων τομέων έτσι ώστε να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ταυτόχρονα θα εξοικονομήσουμε και μεγάλα ποσά. Και θα βελτιώσουμε και την καινοτομία. η αυτοί που χρησιμοποιούν τις προφέρειες θα είναι πιο αποτελεσματικοί ε, και οι πολίτες θα είναι πιο ασφαλείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει συντάξει γνωμοδότηση και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Σίμονς που θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση της ε, ΕΟΚΕ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, κύριε Πρόεδρε, Ολλανδικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη λοιπόν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν έχουμε ακόμα αναφερθεί στο ζήτημα εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά πάνω σε αυτά που μας είπε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρέπει να πω ότι η ανακοίνωση είναι λογική συνέχεια των προσπαθειών που κατεβλήθησαν όσον αφορά την αποτελεσματικότητά μας και την ενίσχυση της στρατηγικής ελέγχου των θαλασσών. Αυτό αποτελεί τμήμα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τον έλεγχο των θαλασσών. Μπορούμε να τονίσουμε την προστασία, την ασφάλεια, την οικονομία, την προστασία και του περιβάλλοντος στο μέλλον. Εξάλλου, η ανακοίνωση αυτή του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει και αναπτύσσει τη σημασία που έχει η των θαλασσών και την ανταλλαγή πληροφοριών είναι από τα βασικά στοιχεία για την ασφάλεια των θαλασσών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να αναλύσουμε την όλη προβληματική. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει κάποια πράγματα πώς τα κράτη-μέλη θα βοηθηθούν όσον αφορά τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού τους χωρίς συμπληρωματικούς πόρους διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μείωση των οικονομικών πόρων. Εξάλλου, γνωρίζει η Επιτροπή ότι χρειάζονται οικονομίες και ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να επενδύσουμε τις οικονομίες μας στη γενική βελτίωση των συστημάτων και στη σωστή εφαρμογή του ΣΥΖΕ. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, τα στερεότυπα, τις νοτροπίες, τις διαδικασίες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να αναλυφθούν πρωτοβουλίες, κυρίως όσον αφορά την κατάρτιση και την ενημέρωση. Θα πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη που υπάρχει όσον αφορά την χρήση των υφισταμένων μηχανημάτων και συστημάτων. Θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών όπως το Φόρουμ των Ακτοφυλακών του Βόρειου Ατλαντικού να γίνεται γενικά μια ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει στη διάθεση όλα τα μέσα που θα επιτρέψουν να ξεπεραστούν τα πολιτισμικά και τεχνικά εμπόδια. Να διευκολυνθεί η εφαρμογή της πρωτοβουλίας. ΣΥΣΕ. Εξάλλου κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών, των πληροφοριών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις διάφορες απειλές που ίσως φανούν. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στον τομέα της ασφάλειας αυτές τις πτυχές. Για τα λιμάνια, για τους εξοπλισμούς κλπ. και για τα φορτία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπώς να λάβει υπόψη επίσης την ασφάλεια του χώρου σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών και να κάνει ό,τι πρέπει στα πλαίσια του ΣΥΣΕ. Η έκθεση του 2013 που παραψιάστηκε από το Office Accountability των ΗΠΑ και παρουσιάζει διάφορες υποδομές που υπάρχουν, επιμένει επί του κατεπήγοντος χαρακτήρα της όλης καταστάσεως. Την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι στη Ουάσιγκτον συζητήθηκε ξανά το θέμα. Ιδού κύριε Πρόεδρε, οι γενικές γραμμές της γνωμοδοτήσεως που θέλουμε να εκφράσουμε ένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και στην Επιτροπή σας και στον εισηγητή σας και στις 24 Μαρτίου ε, διοργανώνει μια διάσκεψη για τις ασφαλείς θάλασσες, Safe Sea, η Επιτροπή μας και θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Keith Taylor έχει το λόγο. Όχι, ο Βιμ Βάντεκαμπ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις πολύτιμες αυτές πληροφορίες που ακούστηκαν. Ελπίζουμε να λάβουμε και αντίγραφο αυτής της ε, παρουσίασης για να την έχουμε και εμείς στο αρχείο μας. Ομολογώ ότι ανησυχώ 400 υπηρεσίες στην Ευρώπη ασχολούνται με την προστασία και την ασφάλεια στη θάλασσα, αν κατάλαβα σωστά. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις ΙΠΑ όπου ε, έχουν μία και μόνο υπηρεσία που αντιστοιχεί στις 400 δικές μας και το ερώτημα είναι βρισκόμαστε ως Ευρώπη στο σωστό δρόμο. Αυτό που με εντυπωσίασε στην ε, παρουσίασή σας ήταν ο όρος εθελοντικός και στη συνέχεια το τι δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πού βρίσκεται τελικά η συνεργασία. Αφενό, θα μπορούσε κανεί να συγχωνεύσει όλε αυτέ τι υπηρεσίε και να δημιουργήσει μία και μοναδική. Και από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε ε, να υπάρξει ένα σύστημα όπου η συνεργασία θα ήταν ε, ε, εθελοντική, προαιρετική. Μήπως θα μπορούσαμε όμως να έχουμε μια πιο δομημένη μορφή συνεργασίας με περισσότερα κίνητρα. Γιατί το να υπάρχουν 400 υπηρεσίες είναι υπερβολή νομίζω. Ε, είχαμε πριν από λίγο καιρό παρακολουθήσει μία ε, παρουσίαση για το Costa Concordia. Ποια είναι ε, η σύνδεση μεταξύ του ατυχήματος αυτού και του CISE και στη συνέχεια τι σχέση έχει το CISE με τους ετούντες άσυλο. Ίσως θα μπορούσε αυτό το σύστημα να βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν τις καταστροφές στη θάλασσα, έχουμε το ζήτημα της ε, Μεσογείου, ε, τα ατυχήματα και αφενός και αφετέρου τα, τα ζητήματα της ε, Μεσογείου και τους ετούντες άσυλο. Ευχαριστώ για τη χρήσιμη αυτή η παρουσίαση. και εγώ έθεσα το θέμα του τραγικού ατυχήματος του και περιμένουμε ακόμα απάντηση. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν ζητήματα για το ποιος ε, ε, επιβαίνει στα πλοία και κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι που ασκούνται, ακόμα και αν θεωρητικά υπάρχουν διαδικασίες. Και οι πληροφορίες δεν μοιράζονται με τον δεδειγμένο τρόπο. Και είχα συγκεκριμένη ερώτηση. Έχουμε μεγάλο εργατικό δυναμικό στον τομέα ναυτιλίας, 600.000 ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ναύτες, τα συνδικάτα και οι κοινωνικοί εταίρες κατά πόσο εμπλέκονται στις συνομιλίες, δηλαδή για το πώς η θαλάσσια εποπτεία θα διεξάγεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ, Keith το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είχα δύο ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θα μπορούσε να παρουσιάσει λεπτομέρειες όσον αφορά τη συνεργασία με το στατιωτικό τομέα και το στατιωτικό έλεγχο. Νομίζω ότι αναφέρθηκε στα πλαίσια του ελέγχου των συνόρων. Το έθεσα αυτό το ερώτημα στα πλαίσια της διαφάνειας. Δεύτερο ερώτημα. Απέτυχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τα συμπληρωματικά καθήκοντα που υπερψήφισε η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο που θα έπρεπε να ανατεθούν στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών όσον αφορά την εποπτεία ε, και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων των υπερακτίων για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Τι εχέγγυα μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΕΜΣΑ όσον αφορά την εκτέλεση των νέων ρόλων που της έχουν αντεθεί. Ευχαριστώ η κυρία Γκμίντα από την ε, Επιτροπή για να απαντήσει στα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια θα συνεχίσω στα αγγλικά. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για μένα γιατί πάντα δουλεύουμε στα αγγλικά. Να ξεκινήσω με τα οικονομικά με τη χρηματοδότηση. Ένα τέτοιο σχέδιο διαλειτουργικότητας προφανώς κοστίζει. Κάναμε μια μελέτη και έχουμε κάποια νούμερα, αλλά είναι δύσκολο κανείς να τα σταθμίσει σωστά γιατί βασιζόμαστε στα στοιχεία τα που μας δίνουν τα κράτη-μέλη, πρόκειται για εθνικές αρμοδιότητες. Πάντως ε, το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από τα ωφέλη που θα προκύψουν, γιατί ε, αν το δείτε το κόστος, για κόστος ενός ευρώ η εξοικονόμηση που θα γίνει θα είναι 9 ευρώ. Ένα προς 9 λοιπόν. Η γνωμοδότησή σας είναι πάρα πολύ καλή και θα είναι πολύ χρήσιμη το είδαμε και στην ε, συνάντηση που οργάνωσε η ΟΚΕ. Πάντως είναι σαφές ότι αν τα κράτη-μέλη θελήσουν να εξυγχρονίσουν τα συστήματά τους με ε, πόρους του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, αυτό μπορεί να γίνει. Υπάρχει δηλαδή κάποια μικρή, μικρή δυνατότητα ενίσχυσης. Ο κύριος Τέιλορ μίλησε για τη χρήση της, ε, τη, τη χρηματοδότηση της ΕΜΣΑ για ε, εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ε, το project αυτό δεν αφορά ένα μόνο τομέα. Ε, θέλουμε με διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριών που υπάρχουν για όλους τους τομείς. Συνεπώς η ΕΜΣΑ προφανώς θα θα συμμετάσχει, μάλλον ο ΕΜΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφαλεία στη Θάλασσα, ε, και θα ωφεληθεί κιόλα, διότι θα πάρει και περισσότερες πληροφορίες. Οπότε, ο, ο ΕΜΣΑ ήδη έχει τέσσερις ε, πλατφόρμες επιτήρησης των εξορρυκτικών δραστηριοτήτων και μπορεί να ωφεληθεί ακόμα περισσότερο μέσω της ε, ε, πρόσβασης σε περισσότερες πληροφορίες που θα εξασφαλιστεί με αυτό το μηχανισμό. Τώρα, για το θέμα της εκπαίδευσης. Πολύ καλή παρατήρηση. Η καινούρια γενιά πληροφοριακών συστημάτων και το ΣΥΣΕ e δεν είναι πληροφοριακό σύστημα, απλά ε, ενώνει πληροφοριακά συστήματα έτσι ώστε να μπορούν να μιλούν μεταξύ τους, να το πω έτσι απλά. Ε, θα χρειαστεί λοιπόν μια καινούργια γενιά πιο κατερτισμένων ε, ελεγκτών και επιτηρητών και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε υπάρχουν τα δίκτυα κατάρτισης γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση για τις ΗΠΑ. Έχω πάει στις ΗΠΑ και στην ακτοφυλακή των ΗΠΑ και όλοι ε, με κοιτούν και ζαλίζονται. Ε, μου λένε <laughs> είστε σίγουροι ότι κάνετε το σωστό στην Ευρώπη. Αυτοί έχουν το μίσε, εμεί έχουμε το ΣΥΣΕ, αυτοί έχουν το μίσε, Maritime Information Sharing Environment, έχουν παρόμοια προβλήματα με εμά που έχουν περισσότερο σχέση με νοοτροπία, με την νοοτροπία της συνεργασίας, με την, ε, διότι ακόμα και στη μία ενιαία ακτοφυλακή υπάρχουν πολλά διαφορετικά τμήματα, αντιλαμβάνονται βέβαια περισσότερο ότι το δικό μας έργο είναι πιο συσήφιο από το δικό τους. 400, 400 φορείς είναι ένα ωραίο νούμερο, το χρησιμοποιώ, ε, όμως και στα κράτη-μέλη μπορούν να γίνουν προσπάθειες να συνεργαστούν μεταξύ τους οι εθνικές αρχές. Και το ΣΥΣΕ θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό πνεύμα, μια κοινή νοοτροπία και να εξασφαλιστεί η αλληλοκατανόηση. Ε, τα ευρωπαϊκά δίκτυα του ΕΜΣΑ, της Frontex κλπ. βοηθούν τα κράτη-μέλη σε αυτή την προσπάθεια. και στην Κομισιόν συζητήσαμε επιμακρών το ε, θέμα του εθελοντικού χαρακτήρα. Μιλάμε για τομεί οι οποίοι έχουν, διέπονται από διαφορετική νομοθεσία, από διαφορετικές νομοθεσίες και μια και μιλούμε και για συνέντευξη μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών θα ήταν αδύνατον να εκδώσουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. η στρατιωτική πτυχή δεν μπορεί επουδενή να διέπεται ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης το ίδιο και οι ε, αστυνομικές αρχές. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και πιο κλασικούς τομείς, ο οποίους μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε επιλέξει αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Υπάρχουν κίνητρα, διότι η βελτίωση της ε, αποτελεσματικότητας είναι ε, απολύτως απαραίτητη σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν όλο και λιγότερα κονδύλια διαθέσιμα. Οπότε λοιπόν αυτή η ανάγκη αποτελεί και κίνητρο. Σε ατυχήματα όπως του Κώστα Κονκόρδια όλοι παρευρίσκονται, όλοι βοηθούν. Δεν θέλω να ε, κρίνω το πώς ε, τη χειρισμού έτυχε το ατύχημα αυτό, δεν είμαι ειδική, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλοι βοήθησαν, κανένας δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να προβλέψει ένα τέτοιο ατύχημα μέσω ενός κοινού συστήματος ε, πληροφοριών. Όμως, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει στην, στον εντοπισμό συγκεκριμένων ε, ε, ροών μετανάστευσης διότι κάθε χώρα έχει το, τους δικούς μηχανισμούς, πολιτικούς μηχανισμούς που ξεκινούν να λειτουργούν μέσα στα σύνορα τους. Αντίθετα, ο στρατός ε, δραστηριοποιείται και εκτός των σύνορων στην ανοιχτή θάλασσα, οπότε θα μπορούσε μια συνεργασία να βοηθήσει. Οι πολιτικές με τις στρατιωτικές αρχές, οι πολιτικοί με τους στρατιωτικούς φορείς θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να ε, προλάβουμε και ατυχήματα στην ανοιχτή θάλασσα. Το project ε, δεν προβλέπει συνεργούς ελέγχους από το στρατό, ε, που ε, Δεν έχουμε στόχο να εξαιρεστούμε καινούρια νομοθεσία, ούτε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων φορέων αυτή τη στιγμή. Όμως, ορισμένα καθήκοντα του στρατού θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολιτικούς φορείς. Για παράδειγμα στην Γαλλία ο στρατός μπορεί να ε, αναλάβει ευθύνες της ακτοφυλακής και οι ευθύνες άλλων πολιτικών φορέων, μη στρατιωτικών φορέων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συνδικάτα, δεν έχω να πω και πολλά πράγματα, διότι πρόκειται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημοσίων φορέων κρατικών φορέων. Καλό θα ήταν να συζητήσουμε το πώς γίνεται η επιτήρηση της ε, θάλασσας και πιστεύω θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ. Έκανα ένα λάθος. Δεν έδωσα το λόγο στην ε, Κλάουντιο Μοντέρο, αλλά θα της τον δώσω τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που με σκεφτήκατε που με θυμηθήκατε τελικά. Ευχαριστώ πολύ την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση. Η, στρατη, η, θαλάσσια, η γαλάζια θαλάσσια στρατηγική και η στρατηγική επιτήρηση του Ατλαντικού ωκεανού δείχνουν ότι η Ευρώπη κοιτάει προς τη θάλασσα θάλασσα που πολλές φορές ε, μας διχάζει αλλά τις περισσότερες φορές μας ενώνει. Και χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτάει πιο μακριά από τις παραδοσιακές δραστηριότητες. Είναι πολύ καλή λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, θα γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή των στόχων της κοινή θαλάσσιας πολιτικής. Το πρόγραμμα ΣΥΖΕ ε, προβλέπει την, προβλέπει την συμμετοχή τρίτων χωρών και αν όχι δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να διευρύνουν το σύστημα αυτό και ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί οι κίνδυνοι δεν σταματούν στα σύνορά μας. Πώς ε, συμμετέχει ο ΕΜΣΑ ε, και πώς συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο στις, στα καθήκοντά του. Τρίτον, ένα από τα εμπόδια είναι η εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών. Πώς πιστεύει η Κομισιόν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ε, αυτού του είδους τα εσωτερικά προβλήματα οργάνωσης των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μία πρόσθετη ερώτηση. Θυμάμαι τον Βίλι Πίτσικ που ήταν μέλος της Επιτροπής μας για πάρα πολλά χρόνια και έλεγε πάντοτε ότι στην Γερμανία ο, εξωτερικός, ε, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και ο Υπουργός ε, ε, Οικονομικών είναι υπεύθυνοι, είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια στη θάλασσα. Αν συνυπολογίσει κανείς και τα 16 κρατήδια τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται και ήταν πάντοτε το κρατήδιο της Ηλεσίας ε, εκείνο που ε, υποστήριζε τη δημιουργία μίας και ενιαίας ε, αρχής για την επιτήρηση της ασφάλισης στη θάλασσα. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε και κάτι με αφορμή αυτό. Για τις τρίτες χώρες. Δεν συμμετέχουν διότι τα κράτη-μέλη σαφώς θέλανε να παραμείνει για αυτά και τις χώρες ΕΟΧ. Έχουμε πολύ ενεργό συμμετοχή της Νορβηγίας στο το πρόγραμμα, διότι έχουν και μεγάλη εμπειρία από τη θάλασσα Μπάρεντς, αλλά μέχρι τώρα δεν συμμετέχουν άλλες τρίτες χώρες, διότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ήδη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα καταστήσει ανέφικτο το εγχείρημα. Τούτο ελεγχθέντος η Ευρωπαϊκή ε, στρατηγική για την ασφάλεια των θαλασσών που θετήθηκε το Συμβούλιο έχει μεγάλη συνιστόσα όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, αναβάθμιση, στήριξη των τρίτων χωρών ε, για την προσπάθεια εποπτείας των θαλασσών, να τους βοηθήσουμε να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την επίτευξη παρομοίων στόχων. Όσον αφορά τις ε, δομές, σαφώς δεν αναφερθήκαμε στις δομές, κυρίως όχι στην ανακοίνωση που σας παρουσίασα, διότι είναι προνόμιο εθνικό και αρμοδιότητα κάθε κράτο κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίζει επί των δομών για τον έλεγχο των θαλασσών. Όμως μπορώ να πω με το παράδειγμα του κυρίου Κράμερ ότι υπάρχει κάποια μετακίνηση προς παρόμοια συστήματα, το πούμε έτσι. Και αυτή η μετακίνηση κινητοποιείται μέρη από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσης όπως τη Eurosurvey, όπου έχεις ένα εθνικό κέντρο συντονισμού για το Eurosur για την εφαρμογή του Eurosur για την ασφάλεια των συνόρων, όπου εκεί και άλλες αρχές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν αν το επιθυμούν και αποφάσισαν πολλά κράτη-μέλη ότι θα ήθελαν και άλλες αρχές να συμμετάσχουν. Παραδείγματο χάρη, αν δείτε τι γίνεται στη Γερμανία, στο Wilhelmshaven, Cuxhaven μάλλον, κατασκευάζουν ένα κέντρο για πληροφορίες για τις θάλασσες και 7 φορείς ε, οι αρμόδιοι είναι παρόντες ήδη υπάρχει κάποια υποδομή, ετοιμάζουν νέο κτίριο για το μέλλον και αυτό το πρότυπο κοινού χώρου συνεργασίας είναι κάτι που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Πιθανότατα είναι η πιο περίπλοκη εκδοχή του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού για τις θάλασσες. Το είδα στην Ολλανδία, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που ακολουθούν παρόμοια κίνηση όσον αφορά ε, κοινή τοποθέτηση σε κτίριο των διαφόρων φορέων. Κάθε αρχή πρέπει να έχει δικό της νομικό σύστημα και όλοι θα πρέπει να σέβονται τα νομοθετικά όρια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να σχεδιαστεί βάση εθνικής νομοθεσίας διότι η εθνική νομοθεσία και συνταγματικό πλαίσιο ε, καθορίζει τις δυνατότητες των εποπτικών φορέων. Ελπίζω έτσι να διευκρινίζω τα πράγματα. Είναι ένα θέμα όπου θα ήταν καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να το συζητά και η επιρροή σας ε, μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ευκαιρίες συνεργασίας. Μαζί τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα και υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα της ενέργεια διάταξη και ε, ε, πάμε στο επόμενο θέμα, ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων και αυτό το θέμα θα συζητηθεί και κλεισμένο των θερών, αλλά μπορούν τα μέλη της Επιτροπής να παραμείνουν εδώ. Δεν είναι όμως δημόσιες. Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω όσοι δεν είναι ευρωβουλευτέ, δεν είναι μέλη της Επιτροπής, να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Θα κάνουμε και ένα διάλειμμα 2-3 λεπτών.